Καλωσορίσατε στη συνεδρία της Επιτροπής Προπολογισμών. Καθίστε σας παρακαλώ πολύ. Το πρώτο σημείο στην ημερήσια διάταξη συνήθω είναι η έγκριση της ημερήσιας διάταξης. Αν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις μπορούμε να την εγκρίνουμε. Δεύτερο σημείο, ανακοινώσεις του Πρόεδρου. Οι αποφάσει των ιστών τη συνεδρίας της 3 Σεπτεμβρίου 2019 είναι διαθέσιμε στον φάκελο τη συνεδρίασης και αν δεν υπάρχουν αντιρρήσει, οι αποφάσει αυτέ μπορούν να θεωρηθούν ότι είναι εγκεκριμένε. Τρίτο σημείο, έγκριση των πρακτικών. Πάλι, αν δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, προσέξτε μας παρακαλώ πολύ. Θεωρώ ότι εγκρίνονται και τα πρακτικά της συνεδρίασης της 3 Σεπτεμβρίου 2019. Τώρα περνάμε στο σημείο 4. Ώρα ψηφοφορία. Σημείο 4. Ψηφοφορία και το προπολογισμό 2019 τμήμα 3. Αιτήσει μεταφορά. Δεν υπάρχουν εδώ αιτήσει μεταφορά. Δεν έχουμε λάβει κάποια τέτοια αίτηση. Άρα μπορούμε να περάσουμε αμέσω στο σημείο 5. Προπολογισμό 2019 άλλα τμήματα και σχετικέ μεταφορέ. Το λόγο κανονικά εδώ πέρα θα έπαιρνε ο κύριος Φερνάντες, ο οποίος είχε αποχωρήσει όμως από την αίθουσα. Θα τον αντικαταστήσει κάποιος, θα πάρει κάποιος το λόγο για το σημείο αυτό. Αν όχι να δώσω το λόγο στους κοιόδης συγητές ενδεχομένω. Φαντάζομαι ότι δεν υπάρχει καμία αντίρρηση, όλοι μου χαμογελάτε από ό,τι βλέπω, μπορούμε να εγκρίνουμε και τις προτινόμενες εδώ μεταφορές, συμφωνείτε. Ευχαριστώ πολύ. Ανά και ο Φερνάντες. Αναφερόμενο στο σημείο 5 της ημερήσιας διάταξης όσον αφορά τις αιτήσει μεταφοράς για τον προπολογισμό του 2019, άλλα τμήματα, πέρα από το τμήμα 3 δηλαδή. Σας ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε η μόνη μεταφορά που έχουμε εδώ πέρα για την οποία δεν υπάρχει πρόβλημα και ας μιλήσω και την ε, μητρική μου γλώσσα, τα πορτογαλικά. Το μόνο σημείο εδώ πέρα που έχουμε ως αίτηση μεταφοράς είναι για το άρθρο 103 και το άρθρο 231. Όσον αφορά το άρθρο 231, αυτό αφορά τη μετάφραση και έχει να κάνει με μια μεταφορά 15.000 ευρώ. Το ποσό αυτό θα αντικατασταθεί από τις εξοικονομήσεις ουσιαστικά που έχουν γίνει στο άρθρο 103 για το Ταμείο Συντάξεων. Έχουμε ακόμα μια αίτηση μεταφοράς. Μάλλον δεν υπάρχουν άλλες αιτήσει μεταφοράς. Απλώς ήθελα να σας πω ότι είμαι υπέρ των δύο αυτών αιτήσεων, κύριε Πρόεδρε όσον αφορά τις γραμμές αυτές του προπολογισμού, Ombudsman 5 κάθετος 2019, Ευρωπαίος Διαμεσολαβητής δηλαδή. Σας ευχαριστούμε πολύ. Θέλει να πάρει κάποιος το λόγο μετά τον κύριο Φερνάντε για το ζήτημα αυτό. Αν όχι, ας επαναλάβω αυτά που είπα πριν από λίγο. Αν δεν υπάρχουν περαιτέρω αντιρρήσεις, οι συγκεκριμένε αυτές αιτήσεις μεταφοράς εγκρίνονται. Σας ευχαριστώ πολύ. Περνάμε στο σημείο 6 της σα διάταξης, κτηριακή πολιτική, Πάλι εδώ πέρα δεν υπάρχει κάποιο συγκεκριμένο ζήτημα στην ημερήσια διάταξη το οποίο πρέπει να εξετάσουμε. Πολύ ωραία. Περνάμε έτσι στο σημείο 7 της ημερήσιας διάταξης. Μάλλον εκτός αν η κυρία Φαμπιάν Κέλλερ θέλει να πάρει το λόγο. Όχι. Πολύ ωραία. Σημείο 7 λοιπόν της ημερήσιας διάταξης, παρουσία του σχεδίου έκτακτης ανάγκης για το Brexit. Δεν έχει έρθει όμως ο ο κύριος Κόπμαν, ο οποίο θα έκανε την παρουσίαση για το σημείο αυτό. Μπορούμε να πούμε στο σημείο 8 τότε. Κρύβεται κάπου μήπως. Λοιπόν, να περάσουμε τότε στο σημείο 8 τη ημερήσια διάταξη. Γενικό Προπολογισμό Ευρωπαϊκή Ένωση για το Οικονομικό Έτο 2020. y a Ah oui La semaine passée. Je, je l'ai rencontré So, yeah, the Commission has proposed a Brexit Ήρθε όμως ο μιλητής. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει προτείνει μέτρα έκτακτη ανάγκη όσον αφορά το Brexit για τον προπολογισμό 2020, ακολουθώντα μια ανάλογη πρόταση που είχε γίνει για τον προπολογισμό 2019. Προβλέπεται εδώ πέρα η διαδικασία σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Η σύμφωνη γνώμη θα πρέπει όμω να υποβληθεί σε σχέση με το σχέδιο απόφαση του Συμβουλίου. Το Συμβούλιο έχει αρχίσει να επεξεργάζεται την πρόταση αυτή. Οι συντονιστέ αποφάσισαν να αναλάβω εγώ το φάκελο αυτό ως πρόεδρος της Επιτροπής Προπολογισμών, όπως κάτι ανάλογο είχε κάνει ο προηγούμενος πρόεδρος για το σχέδιο προπολογισμού 2019. Εύχομαι βέβαια το Ηνωμένο Βασίλειο να μην αποχωρήσει χωρίς συμφωνία, αλλά θα πρέπει να προετοιμαστούμε και για το δεχόμενο αυτό. Είναι πολύ σημαντικό να ασχοληθούμε γρήγορα και εγκαίρω με το ζήτημα αυτό, καθότι είναι πιθανό το Ηνωμένο Βασίλειο να αποχωρήσει χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Δίνω λοιπόν ευθύ αμέσω το λόγο στον κύριο Κόπμαν, ο οποίο είναι Γενικό Διευθυντή τη Γενική Διεύθυνση Προπολογισμού τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή, προκειμένου να μα παρουσιάσει την πρόταση τη Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Κύριε Κόπμαν, έχετε το λόγο. Σα ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Καλημέρα σε όλου. Δράτω με τις ευκαιρία προκειμένου να σα παρουσιάσω το σχέδιο αυτό έκτακτης ανάγκης και το σχετικό κανονισμό σε περίπτωση που έχουμε τελικά Brexit χωρίς συμφωνία, μήπως θα μπορούσαμε να δούμε και τις διαφάνειες τις οποίες έχουμε ετοιμάσει. Να ξεκινήσω λέγοντας ότι η πρόταση αυτή αποτελεί τμήμα μιας δέσμης μέτρων, η οποία εγκρίθηκε στις 4 Σεπτεμβρίου Και στην ουσία, στόχος τη θέσμη αυτή μέτρων είναι να δώσει στον Ομένο Βασίλειο τη δυνατότητα να συνεχίσει να συμμετέχει στον προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ακόμα και αν δεν υπάρξει τελικά συμφωνία σε σχέση με το Brexit. Προβλέπεται δηλαδή να συνεχιστεί η επιλεξιμότητα του Ηνωμένου Βασίλειου και των σχετικών δικαιούχων στα προγράμματα δαπανών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και βέβαια θα πρέπει εδώ πέρα το σχετικό αυτό πρόγραμμα να προσαρμοστεί στις ε, προϋποθέσεις, του όρους που ισχύουν στα πλαίσια του ενωσιακού δικαίου και αυτό μπορείτε να το δείτε μάλιστα στο σχετικό κανονισμό 2019 κάθετος 1197, ένας κανονισμός που άρχισε να ισχύει νωρίτερα φέτος. Όσον αφορά τώρα τους βασικούς στόχους της πρότασης αυτής, πρέπει να είμαι ιδιαίτερα σαφής, δεν ξέρω αν μπορείτε να δείτε τώρα και τις διαφάνειες. Ο βασικός στόχος της πρότασης αυτής είναι διτός. Αφενός θέλουμε να έχουμε μια συντεταγμένη έφτακτη εφαρμογή και εκτέλεση του προπολογισμού και αφετέρου. Θέλουμε επίσης να μετριάσουμε πιθανούς κλειδονισμούς πιθανή αναστάτωση που θα μπορούσε να προκύψει για τους δικαιούχους του Ηνωμένου Βασιλείου ή ακόμα και για δικαιούχους εκτός Ηνωμένου Βασιλείου, δηλαδή από τις υπόλοιπες 27 χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης που ενδεχομένω να συμμετέχουν σε κοινά προγράμματα με το Ηνωμένο Βασίλειο όσον αφορά για παράδειγμα το τομέα της έρευνας ή άλλους τομείς. Τώρα, τα βασικά στοιχεία της συγκεκριμένη πρότασης ε, δεν θα σας κάνουν ιδιαίτερη εντύπωση, δεν υπάρχει κάποια καινοτομία εδώ πέρα. Ακολουθούμε τις συνήθεις βασικές μας αρχές και τη βασική δομή και διάρθρωση που έχουμε σε σχέση με τον υφιστάμενο κανονισμό του Συμβουλίου 2019-1197, ε, όπου προβλέπεται ένα πλαίσιο έκτακτη ανάγκης ε, για το έτος 2019. Προσπαθούμε να κάνουμε ελάχιστες προσαρμογές, αντιγράφοντας ουσιαστικά τις βασικές διατάξεις που έχουν εγκριθεί για το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης για τον προπολογισμό του 2019 και όπω και στο πλαίσιο έκτακτη ανάγκη του 2019, έτσι και στο εφιστάμενο πλαίσιο προβλέπεται ότι κανένα κράτος μέλος δεν θα πρέπει να επιβαρυνθεί περισσότερο, δηλαδή δημοσιονομική ουδετερότητα για τα 27 κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης πέρα από το Μένο Βασίλειο. Αυτό προσπαθούμε να το διαφυλάξουμε πάση θυσία. Και έπειτα, το ποσό το οποίο θα πρέπει να καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο προφανώς έχει να κάνει με το συνολικό μερίδιο ιδίων πόρων σε σχέση με το σχέδιο προπολογισμού του 2020, αλλά βέβαια και εδώ πέρα θα πρέπει να γίνει μια σχετική προσαρμογή, λαμβάνοντας υπόψη και τις συνολικές δαπάνες που θα εγκριθούν τελικά στο πλαίσιο του προπολογισμού για το 2020. Εδώ πέρα θα πρέπει να, έχουμε, να κάνουμε κάποιες προσαρμογές σε σχέση με το 2019. Προτείνουμε τώρα και ένα χρονοδιάγραμμα λίγο διαφορετικό σε σχέση με το χρονοδιάγραμμα το οποίο προτάθηκε για το προηγούμενο πλαίσιο έκτακτης ανάγκης. Ζητάμε προκειμένου από το Ηνωμένο Βασίλειο την 1η Ιανουαρίου του 2020, μέσα σε 7 ημερολογικές μέρες μετά τη θέση ενισχύ του κανονισμού αυτού, να υποβάλει μια γραπτή δέσμευση ότι όντως πληρεί όλες τις προποθέσεις και όλους τους όρους του σχετικού κανονισμού και ότι επομένως το Ηνωμένο Βασίλειο πρόκειται να χρησιμοποιήσει τη δυνατότητα που του δίνει ο νέος αυτός κανονισμός σε σχέση με τη δυνατότητα χρηματοδότησης και κάτι που είναι πολύ σημαντικό το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να δεχθεί όχι μόνο τη χρηματοδότηση βέβαια της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά και τους ελέγχους και τις επιθεωρήσεις που κάνουν τα αρμόδια όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και εν συνεχεία, το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να καταβάλει την πρώτη πληρωμή στις 20 Ιανουαρίου ή 20 ημερολογιακές μέρες μετά τη θέση ενισχύ του εν λόγω κανονισμού. Ουσιαστικά αυτό θα αντιστοιχεί σε ποσό τριών μηνών. Τώρα, όσον αφορά τα επόμενα βήματα, η προβλεπόμενη διαδικασία εφαρμογή του κανονισμού αυτού ουσιαστικά είναι ταυτόσιμη με την προηγούμενη διαδικασία. Ομοφωνία του Συμβουλίου απαιτείται εδώ. Θα πρέπει να έχουμε έπειτα τη σύμφωνη γνώμη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Είναι πολύ σημαντικό επίσης να σημειώσουμε ότι τόσο η Γερμανία όσο και η Δημοκρατία της Τσεχίας έχουν συγκεκριμένε εθνικέ απαιτήσει όσον αφορά τη σύμφωνη γνώμη την κοινοβουλευτική που πρέπει να δοθεί από τι χώρε αυτέ. Αυτό λοιπόν θα απαιτήσει λίγο περισσότερο χρόνο, αλλά αυτό προβλέπεται ούτω ή άλλω στο σταγματικό του δίκαιο, άρα δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι γι' αυτό. Επομένω, η γρήγορη έγκριση του συγκεκριμένου αυτού κανονισμού είναι πάρα πολύ σημαντική, προκειμένου ο κανονισμό να είναι διαθέσιμο, να μπορεί να εφαρμοστεί και να υπάρχει και ένα πλαίσιο προβλεψιμότητος για τους δικαιούχους και προκειμένου να μπορέσουμε ως Ευρωπαϊκή Ένωση να συνεχίσουμε να εφαρμόζουμε τα όσα προβλέπονται στο πλαίσιο του προπολογισμού για το 2020. Αυτά είναι συντομία όσον αφορά το περιεχόμενο του νέου αυτοκανονισμού. Όπω σα είπα, στα περισσότερα σημεία του ταυτίζεται με τον προηγούμενο κανονισμό και ελπίζω ότι θα καταφέρει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπω είχε εγκρίνει το προηγούμενο πλαίσιο τη ανάγκη, να εγκρίνει και αυτό το πλαίσιο τη ανάγκη που είχε να κάνει με τον προπολογισμό του 2020. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόπμαν. Την επόμενη φορά που θα έρθει να μας κάνετε μια ανάλογη παρουσίαση θα θέλαμε πάρα πολύ να έχουμε εκ των προτέρων τις διαφάνειες προκειμένου να μπορούμε να τις διαβάσουμε και εμείς εκ των προτέρων και να μπορούμε να προετοιμάσουμε παρατηρήσεις και ερωτήσεις. Δεν ξέρω αν θα ήθελα να πάρει κάποιο το λόγο για τυχόν ερωτήσεις κύριε Λόου. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ως επιχειρηματίας ε, πραγματικά εκπλήσωμαι που δεν υπάρχει πληρέστερη εικόνα των συνεπειών της αποχώρησης του Ηνωμένου Βασιλείου χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου. Είναι 50-50 η κατάσταση. Όταν συναντήθηκα με τον κύριο Μπαρνιέ στο Στρασβούργο την περασμένη εβδομάδα, είπα ότι δεν θα υπέγραφα τη συνθήκη του όπως την αποκαλεί, ακόμα και αν είχα χάσει τον πόλεμο. Ε, πιστεύω λοιπόν ότι είναι καθόλου πιθανό να αποχωρήσουμε χωρί συμφωνία και πραγματικά ως επιχειρηματία εγώ θα περίμενα τουλάχιστον το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ή και η Ευρωπαϊκή Ένωση να έχει δύο προπολογισμού. Έναν αν μείνουμε και έναν αν φύγουμε και ο κύριος Μπαρνιέ θα έπρεπε να γνωρίζει και τις συνέπειες της απαχώρησή μας. Εάν φύγουμε χωρίς συμφωνία θα μείνει ένα τεράστιο κενό ε, στον επιχειρησιακό προλογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και πραγματικά λοιπόν με εκπλήσει το γεγονός ότι δεν έχουμε τις πληροφορίες πρόχειρες. Θα έπρεπε να τις έχουμε όλοι στη διάθεσή μας γιατί αν φύγουμε χωρίς συμφωνία όλοι οι υπόλοιποι θα πρέπει να πληρώσουν πάρα πολύ περισσότερα ε, χρήματα. Ε, η άλλη παρατήρηση είναι ότι αν δούμε την εικόνα της Ευρώπης, την πρόβλεψη η οποία επιδεινώνεται, μήπως θα έπρεπε να κάνουμε περικοπές αντί να αυξάνουμε το συνολικό κόστος. Θεωρώ ότι είναι το σωστό για όλες τις περιφέρειες στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τους πολίτες μας, ιδίω επειδή το ευρώ ε, οδηγεί του περισσότερους στη φτώχεια. Ε, ξέρω ότι προτείνεται να κλείσουμε τα κενά με διάφορες φορολόγηση στα πλαστικά και σε διάφορα άλλα. Πραγματικά όμως αν δούμε τη χρονιά, πραγματικά χρειαζόμαστε δύο προπολογισμού. Έναν να αποχωρήσουμε χωρίς συμφωνία και έναν εάν συνεχίσουμε να πληρώνουμε. Και οι προτάσεις που βλέπω εδώ είναι ότι η, η κλασική περίπτωση της Ευρωπαϊκής Ένωσης που θέλει και την πίτα ολόκληρη και το σκύλο χορτάτο. Πραγματικά ε, θεωρείται ότι είμαστε κράτος παρίας; ε, θα πρέπει να δούμε κάτι περισσότερο, πρέπει ε, να ξεκινήσουμε μάλιστα και σύντομα για να υπάρχει και κάτι ουσιαστικό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Χάουαρτ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Έχω ακούσει ένα σωρό ανοησίες από το κόμμα που είναι υπέρ του Brexit από τότε που ε, επανεξελέγησαν προσφάτως. Ε, οι ανοησίες του κόμματος του Brexit είναι αυτά τα πράγματα τα οποία πραγματικά έχουν βουλιάξει το Ηνωμένο Βασίλειο. Αυτό δεν αφορά το μελλοντικό προπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αφορά τη δυνατότητα των Βρετανικών Ιδρυμάτων που είναι εταίροι σε ευρωπαϊκά προγράμματα να συνεχίσουν να συμμετέχουν σε αυτά τα προγράμματα μέχρι το τέλος του 2020 εάν η Βρετανική κυβέρνηση αποφασίσει ότι αυτό είναι αυτό το οποίο επιθυμεί να κάνει εάν η Βρετανία αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς συμφωνία στις 31 Οκτωβρίου που πραγματικά ελπίζω ότι δεν θα κάνει το καθαρό αποτέλεσμα αποχώρησης χωρίς συμφωνία και όχι να συμμετέχει και στον προπολογισμό, όπως ε, ε, φαίνεται να επιλέγει η Βρετανική κυβέρνηση, που σε καμία περίπτωση δεν είναι η θέση ενός ε, κράτους παρία, θα επιτρέψει στα Βρετανικά πανεπιστήμια να συνεχίσουν να εργάζονται ανενόχλητα στα ευρωπαϊκά ερευνητικά προγράμματα στα οποία συμμετέχουν. Θα επιτρέψει και στην οργάνωση που επισκέφτηκα χθε στο Brighton που ε, παράγει βρετανικές ταινίε με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση και εκπαιδεύει ανθρώπου ε, στη δημιουργική βιομηχανία τη Βρετανία να συνεχίσουν να υποφελούνται από το πρόγραμμα Δημιουργική Ευρώπη. Να υπάρχουν και δυνατότητε ε, για επιδοτήσει σε Βρετανού ε, γεωργούς και φυσικά θα δώσει τη δυνατότητα σε εταίρους εντός Ευρωπαϊκής Ένωσης να συνεχίσουν και αυτοί τη δική τους τη συμμετοχή σε αυτά τα προγράμματα και αυτά τα προγράμματα συνεργασίας είναι προς όφελος όλων. Αυτό λοιπόν σημαίνει ότι θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι θα γίνεται ομαλή μετάβαση χωρίς διαταραχές θέλουμε να εξασφαλίσουμε ότι οι δεσμεύσεις που ανέλαβε το Βρετανικό κράτος θα συνεχιστούν και θα ε, τηρηθούν. Και αυτό θα θέσει τη Βρετανική κυβέρνηση, τη Βρετανικό κράτος σε καλύτερη θέση να δημιουργήσει μια σχέση εμπιστοσύνη με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και αν αυτοί οι ανόητοι πραγματικά ενδιαφέρονται για τη χώρα τους, θα σταματήσουν αυτές τις ηλίφιες ρητορίε και θα κάνουν μια συμφωνία για τη χώρα τους και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Όλμπριχτ. Όλοι θα μιλήσετε με τη σειρά σας ο καθένας. Ε, just, just to ask the Θα ήθελα να ζητήσω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας διευκρινίσει κάτι, διότι αν θυμάμαι καλά τα στοιχεία που μας έδωσε ο Επίτροπος Έτιγκερ πριν από κάποιους μήνες, βάσει αυτών η Βρετανική συνεισφορά, λίγο πολύ, είναι περίπου 17 δις μείον την επιστροφή, δηλαδή κάτι μεταξύ 11 και 12 δις. Αν δεν κάνω λάθος, αυτό είναι το κενό λόγω του Brexit στον ευρωπαϊκό προπολογισμό. 11-12 δις. Από αυτό θυμάμαι ότι ο Επίτροπος μας είχε πει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο παίρνει περίπου 5 με 6 δις το χρόνο. Άρα, δεν θα είναι μείωση 11-12, θα είναι κατά μείον 5 με 6 δις το χρόνο. Επομένως το πρόβλημα του χρόνου για την Ευρωπαϊκή Ένωση, αν τα κατάλαβα καλά, 7, 6-7 δισεκατομμύρια για το 2020. Εάν σταματήσουμε πλήρως, και αυτό είναι για τον κύριο Χάουαρθ, να σταματήσουμε τη χρηματοδότηση των προγραμμάτων στο Ηνωμένο Βασίλειο. Θα υπάρχει πρόβλημα εντό Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή 5 έω 7 δι. Τι γίνεται λοιπόν για τον προπολογισμό του 2020 αν το κενό είναι 5 με 7 δι. Σωστά είναι αυτά που λέω. Γιατί αυτό σημαίνει ότι θα πρέπει να μειώσουμε τον προπολογισμό του 2020 κατά 5 ή ε, έως 7 δις. Για του χρόνου βεβαίως, το κενό για μας, αν θέλουμε να μείνουμε στο ίδιο επίπεδο, θα είναι 12 δις αλλά για το 2020 θα είναι 12 μείον τα βρετανικά προγράμματα. Σωστά, ε, τα υπολογίζω ή κάνω λάθο. Ε, αυτή είναι η ερώτησή μου. Θα ομαδοποιήσουμε τι παρατηρήσει και μετά ο κύριο Κόμπμαν ε, θα απαντήσει ή θα προσπαθήσει τουλάχιστον να απαντήσει. Κυρία Χολμάιερ. Έχω και εγώ μια παρόμοια ερώτηση όπως ο συνάδελφος Όλμπριχτ, αλλά δεν χρειάζεται να σας επαναλάβω την ερώτηση. Για τους συναδέλφους από το Ηνωμένο Βασίλειο που δεν ανήκουν στην ομάδα S&D θα ήθελα να πω ότι δεν νομίζω πως είστε σε θέση να συζητήσετε αυτό το θέμα για, λόγω της πολιτικής. Ευχαριστώ πολύ, κύριος Νίλσεν. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Χόουαρ θα αποτελεί ανόητους ε, τους ε, συμμετέχοντες στο συνέδριο των εργατικών, οι οποίοι βέβαια είχαν μια ξεκάθαρη πολιτική σε ό,τι αφορά τον Brexit. Μετά από ένα καθαρό λοιπόν Brexit, το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα πρέπει να καταβάλει άλλες πληρωμές στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ο κύριο Χόουαρθ μίλησε για τους αγρότες, όμως η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου υποσχέθηκε να αντισταθμίσει τις υφιστάμενε ε, πληρωμές του δικαιούχου στη χώρα. Το θέμα είναι η διασυνοριακή συνεργασία με ε, την ε, μορφή ενώσεων ε, και συνεργασιών με τα πανεπιστήμια και τις επιχειρήσεις. Θα πρέπει λοιπόν οι συνεργασίες αυτές να είναι για πολύ συγκεκριμένα project και η Ευρωπαϊκή Ένωση θα οφείλει να καταβάλει ε, κονδύλια στα πανεπιστήμια του Ηνωμένου Βασιλείου για αυτά τα συγκεκριμένα project. Δεν θα πρέπει λοιπόν να είμαστε επιλεκτικοί και να διαλέγουμε ε, σύμφωνα με τις εθνικές μας προτεραιότητες. Κύριε Χόουαρθ, αυτό ονομάζεται εθνική κυριαρχία και σας προτείνω να κοιτάξετε σε ένα λεξικό. Ευχαριστώ. Κύριε Λαπόρτ. Αν θέλετε να μιλήσετε, παρακαλώ να ζητήσετε το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Αυτή η πρόταση κανονισμού για αποχώρηση χωρίς συμφωνία της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, σημαίνει ότι θα υπάρχει ένα κενό νομικό και πρέπει να βρούμε κάτι ε, για να συμπληρώσουμε αυτό το κενό. Πρέπει οι Βρετανοί δικαιούχοι να είναι επιλέξιμοι δηλαδή για τα ευρωπαϊκά κονδύλια μέχρι το τέλος ε, του 2020 και αυτό σημαίνει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα τηρήσει τι δημοσιονομικέ του δεσμεύσει και θα συμμετέχει στον προπολογισμό τη Ένωση. Μπορεί να διαμορφωθεί διαφορετικά το κείμενο. Μπορούμε να πούμε ότι είναι εντολή προ την Βρετανική κυβέρνηση με αυτή την προσωρινή συμφωνία ή θεωρούμε ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση προσπαθεί να περιορίσει τις, τον αντίκτυπο του Brexit. Το, είτε το επιθυμούν είτε όχι οι Ευρωπαίοι φαίνονται, το Ηνωμένο Βασίλειο θα αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και θα πρέπει λοιπόν να αντισταθμίσουμε λοιπόν τις ε, καθαρές ε, εισφορές ε, που είναι περίπου 12 δις ευρώ. Γιατί να μετατοπίσουμε λοιπόν αυτόν από τώρα με μείωση του ευρωπαϊκού προϋπολογισμού. Ως Γαλλίδα Ευρωβουλευτής θεωρώ ότι η αποχώρηση χωρίς συμφωνία θα έχει αύξηση κατά 1 έως 2 δις ευρώ για μας ως Γαλλία και επομένως για γιατί να έχουμε 150 τροπολογίες τώρα στον προπολογισμό του 2020. Θα πρέπει να ε, δούμε τι θα γίνει. Θα έχουμε 2,7 δις ευρώ παραπάνω σε σχέση με το 2019. Για να ολοκληρώσω θα ήθελα να επιστήσω την προσοχή σας σε κάτι πιο γενικό. Ε, το να σκεφτούμε τις συνέπειες μιας αποχώρησης χωρίς συμφωνία είναι καλή, αλλά θα πρέπει ε, να βρούμε και έναν τρόπο να αποφύγουμε το σκληρό Brexit. Θα πρέπει να δούμε τι θα κάνουμε. Το ψήφισμα που ψηφίστηκε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ολομέλεια ε, δίνει στην Βρετανική κυβέρνηση όλη την ευθύνη για την αποτυχία. Ίσως θα έπρεπε να συζητήσουμε μαζί τους αντί ε, να τους επιρρύπτουμε απλώς ευθύνε. Ο κύριος Παπαδημούλης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Παρακολουθώ με ενδιαφέρον την προσπάθεια να μετατραπεί σε ένα ρίγκ εσωτερικής πολιτικής αντιπαράθεσης στο Ευρωκοινοβούλιο για πράγματα που αφορούν στην εσωτερική πολιτική σκηνή του Ηνωμένου Βασιλείου από μια μικρή ομάδα συναδέλφων, αλλά νομίζω ότι εμείς πρέπει να συγκεντρώσουμε την προσοχή μας σε αυτά που θα απασχολήσουν όσο θα συνεχίσουμε ενωμένοι να δουλεύουμε για το project της Ευρωπαϊκής Ενοποίησης. Και νομίζω ότι είμαστε υποχρεωμένοι να ζητάμε και από την Κομισιόν και από τα κράτη-μέλη ε, εναλλακτικά επεξεργασμένα σενάρια και για τις δύο εκδοχές. Και για το Brexit με συμφωνία και για το Brexit χωρίς συμφωνία. Και θέλω να ρωτήσω την Κομισιόν αν σκοπεύει να αντισταθεί πραγματικά σε μια λογική που κυριαρχεί στο Συμβούλιο δυστυχώς και την οποία το Κοινοβούλιο την απορρίπτει, να αντιμετωπίσουμε το Brexit περικόπτοντας με μια, με μια προσέγγιση business as usual τις δαπάνες για τη συνοχή, τις δαπάνες για την κλιματική αλλαγή, τις δαπάνες για την κοινή αγροτική πολιτική, τις δαπάνες για την πρωτοβουλία για την απασχόληση και τη δημιουργία θέσεων εργασία στην νεολαία. Έχετε σκεφτεί να προτείνετε αύξηση των ιδίων πόρων. Έχετε σκεφτεί να πιέσετε για να αυξηθεί η συμβολή των κρατών μελών. Γιατί θεωρείτε δόγμα ότι μπορούμε να κάνουμε περισσότερα πράγματα με λιγότερα λεφτά, όπως δυστυχώς πιστεύουν ορισμένες κυβερνήσεις. Thank you. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Θα μιλήσω και εγώ τη γλώσσα μου, έτσι ώστε να μιλήσω πιο συγκροτημένα. Οι πράσινοι λοιπόν θεωρούν ότι δεν είναι προς το συμφέρον κανενός να αποχωρήσει το Ηνωμένο Βασίλειο χωρίς συμφωνία και προσωπικά δεν πιστεύω ότι είναι προς το συμφέρον της ίδιας της ε, Μεγάλης Βρετανίας. Ο συνάδελφος από το S&T το παρουσίασε αρκετά σωστά νομίζω. Υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι, πάρα πολλοί οργανισμοί στην ε, Μεγάλη Βρετανία οι οποίοι εποφελούνται. Γι' αυτό χρειάζεται να ε, γίνει κάτι για αυτούς, έτσι ώστε να μην τους αφήσουμε ξεκρέμαστους. Και δεν νομίζω ότι είναι προς το συμφέρον των Βρετανών να μην βρεθεί μια σωστή λύση για την μελλοντική συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Η μη συμφωνία δεν είναι λύση. Κανείς λοιπόν ε, δεν νομίζω ότι μπορεί να υποφεληθεί από αυτό αυτό θα οδηγήσει μόνο σε επιδείνωση της οικονομικής κατάστασης και όχι σε σταθεροποίηση όπως θεωρούν κάποιοι. Οι χρηματοπιστωτικές αγορές νομίζω θα το αποδείξουν. διότι μια άτακτη αποχώρηση του Ηνωμένου Βασιλείου θα κλονίσει την ε, οικονομία όχι μόνο της ε, χώρας αλλά σε παγκόσμιο επίπεδο. Νομίζω ότι είναι προς το δικό μας συμφέρον, προς το συμφέρον της Ευρωπαϊκής ε, Ένωσης ε, να μην ε, κάνουμε περικοπές στα τυφλά από εδώ και από εκεί, έτσι ώστε να εξοικονομήσουμε πόρους. Αυτό θα οδηγήσει στο αντίθετο αποτέλεσμα. Και νομίζω πως υπάρχουν αρκετά προγράμματα τα οποία στηρίζουν πολλές περιφέρειες και γι' αυτό θα έπρεπε να συνεχίσουν να λειτουργούν, να συνεχίσουν οι πληρωμές. Δεν μπορούμε να ακυρώσουμε και να καταργήσουμε προγράμματα έτσι απλά μέσα σε λίγες εβδομάδες. Γι' αυτό λοιπόν ε, θα ήθελα να κάνω μια έκκληση στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή και στο Συμβούλιο να είναι συνετή, να μην ε, υπάρχουν σενάρια τυφλών περικοπών. Αυτό δεν είναι ρεαλιστικό και δεν ανταποκρίνεται στις αξίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης ούτε και στους στόχους της για το κλίμα μεταξύ άλλων. Ευχαριστώ πολύ. Δεν υπάρχουν άλλα σχόλια ή ερωτήσεις. Ο κύριος Πόλοκ. Ευχαριστώ πολύ. Τα θέματα αυτά είναι πάρα πολύ σημαντικά. Όμω έχουν περάσει τρία χρόνια από τότε που το Ηνωμένο Βασίλειο ψήφισε να αποχωρήσει από την Ευρωπαϊκή Ένωση και αυτή η συζήτηση γίνεται ακόμα. Ο Τζον Χόουαρθ μίλησε με προσβλητικά λόγια για τους ευρωβουλευτές του ε, κόμματος Brexit όταν έχουν κερδίσει τις εκλογές με 29 ευρωβουλευτές. Εγώ λέω πως πρέπει να σέβεστε τους ψηφοφόρους, να σέβεστε την ψήφο του Βρετανικού λαού και προς την Ευρωπαϊκή Ένωση λέω ότι πρέπει να σέβονται και εμάς. Είμαστε διατεθειμένοι να κάνουμε μία συζήτηση σχετικά με ε, το πόσα χρήματα πρέπει να καταβληθούν και το τι πρέπει να γίνει, έτσι ώστε να βοηθήσουμε, για παράδειγμα, τα εκπαιδευτικά ιδρύματα να ανταποκριθούν ε, στις ε, υποχρεώσεις τους. Όμως, μην ξεχνάτε, ψηφίσαμε 74 εκατομμύρια ε, άνθρωποι ψήφισαν. Η απόφαση ήταν υπέρ της αποχώρησης και εμείς αυτό περιμένουμε. Σας ευχαριστώ. Ο κύριος ε, Ταμίτζα, να με συγχωρείτε που ήρθα λίγο αργόπορημένος στη συζήτηση αυτή αλλά θεωρώ ότι το Ηνωμένο Βασίλειο είναι μια αρκετά δημοκρατική χώρα. Ε, έχουμε κοινοβουλευτική δημοκρατία και όχι δημοκρατία των δημοψηφισμάτων. Εκτιμώ πάρα πολύ τους συναδέλφους από το κόμμα υπέρ του Brexit. Να πω όμως ότι ένας από τους λόγους που δεν έχουμε αποχωρήσει ακόμα είναι επειδή η συντηρητική κυβέρνηση, η οποία διοργάνωσε το δημοψήφισμα, χρησιμοποίησε το και ενεργοποίησε το άρθρο 50 λίγους μήνες μετά το δημοψήφισμα. Μετά πέρασαν δύο χρόνια μέχρι τις 29 Μαρτίου. Γι' αυτό λοιπόν νομίζω ότι δεν πρέπει να μιλάμε για τρία χρόνια, διότι αυτό ε, δεν είναι σωστό. Τώρα, στο πλαίσιο της κοινοβουλευτικής δημοκρατίας είναι πολύ δύσκολο για την ε, παρούσα κυβέρνηση να ε, κυβερνήσει με μια τόσο μικρή πλειοψηφία. Δεν μπορούν να περάσουν τίποτα από το κοινοβούλιο και αν δεν καταφέρνουν να το κάνουν αυτό στο κοινοβούλιο δεν γίνεται τίποτα. Γι' αυτό δεν ξέρω ποιους άσους έχει στο μανίκι του ο κύριος Τζόνσον, αλλά δεν νομίζω να καταφέρουμε να προχωρήσουμε πριν τις 31 Οκτωβρίου. Ευχαριστώ πολύ. Να υπενθυμίσω σε όλους ότι έχουμε έρθει εδώ για να συζητήσουμε όχι την ε, πολιτική της Βρετανίας, αλλά το ε, θέμα που συζητάμε που έχει να κάνει με το σχέδιο έκτακτης ανάγκης. Γι' αυτό λοιπόν θα περάσουμε στις απαντήσεις. Ε, κυρία Σκέρα μήπως θέλετε να μιλήσετε κι εσείς για βρετανική πολιτική. Όχι. Συμφωνώ απόλυτα με εσάς κύριε Πρόεδρε. Είμαστε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Ηνωμένο Βασίλειο είναι δημοκρατική χώρα η οποία έλαβε μία απόφαση και προσπαθεί να την ε, χειριστεί ως ε, ανεξάρτητη χώρα. Όμως εδώ και 46 χρόνια έχουμε σχέσεις, ε, μας συνδέουν διάφορα προγράμματα κοινά. Μας συνδέει ένας ε, ομφάλιος λόρος με τη Γαλλία, το τούνελ στη Μάνχη. Δεν μπορείτε λοιπόν να ακυρώνετε αυτή την ιστορία τόσο εύκολα μέσω του προπολογισμού. Γι' αυτό λοιπόν θα ήθελα να ρωτήσω τον εισηγητή το εξή. Μας μιλήσατε για τους κινδύνους στην ε, γεωργία, στην έρευνα. Υπάρχουν, ε, υπάρχει κίνδυνο και σε άλλου τομείς σε περίπτωση μη συμφωνίας. Δεδομένη της δυσκολίας εφαρμογής των ευρωπαϊκών ε, προγραμμάτων και πολιτικών. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Κόπμαν. Έχετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Δύο ερωτήσεις ξεχώρισα από την όλη συζήτηση του Όλμπριχτ. Καταρχάς η ερώτηση του κυρίου Όλμπριχτ ε, που μας ρώτησε να αποσαφηνίσουμε τη δημοσιονομική χρηματοοικονομική κατάσταση σε περίπτωση σκληρού Brexit. Νομίζω ότι εδώ πέρα θα πρέπει να κάνουμε μια σαφή διάκριση ανάμεσα σε αυτό το οποίο θέλει να κάνει αυτό το πλαίσιο έκτακτης ανάγκης που στόχος του είναι ουσιαστικά να συνεχίσει να συμβάλλει στον προπολογισμό του 2020 και να μπορεί να αποφεληθεί από τον προπολογισμό αυτό το Νομένο Βασίλειο, η συνεισφορά θα είναι 17 δισεκατομμύρια ευρώ. Αυτό είναι το ποσό που θα πρέπει να καταβάλει το Ηνωμένο Βασίλειο. Βέβαια, το Ηνωμένο Βασίλειο θα λάβει και μία σειρά από ε, ήδη προεγκεκριμένες ε, δαπάνες Επομένως, δεν μπορούμε αυτή τη στιγμή να πούμε ποιες θα είναι οι συγκεκριμένες καθαρές επιπτώσεις όσον αφορά την συνεχιζόμενη συμμετοχή του Ηνωμένου Βασιλείου στο υπερπολογισμό αυτό. Πάντως σε προηγούμενες συζητήσεις είχαμε αποτιμήσει το ποσό αυτό ανάμεσα σε 10 και 15 δισεκατομμύρια ευρώ και νομίζω ότι ε, μπορούμε να συνεχίσουμε με βάση αυτή την εκτίμηση. Πάντως ε, Ο κανονισμός Συμβουλίου για το νέο αυτό πλαίσιο έκτακτης ε, ανάγκης είναι ένα κανονισμό ο οποίος προβλέπει ότι το Ηνωμένο Βασίλειο θα πρέπει να κάνει μια ακαθάριστη ε, συνεισφορά. Τώρα, όσον αφορά τα πλεονεκτήματα της πρότασης αυτής για τους δικαιούχους, τα πλεονεκτήματα αυτά είναι σαφέστατα. Απουσία της, ε, του κανονισμού αυτού και σε περίπτωση αποχώρησης χωρίς συμφωνίας, οι, οι άμεση δικαιούχοι κοινοτικών προγραμμάτων πολύ απλά δεν θα μπορούν πλέον να υποφελούνται από το νέο προπολογισμό σε σχέση με τις πιστώσεις ανάληψη υποχρεώσεων που έχουν προβλεφθεί. Σας ευχαριστούμε κύριε Κόπμαν. Το σχέδιο έκθεσης θα μας απασχολήσει στη συνεδρίαση της 1ης Οκτωβρίου. Θα ψηφίσουμε στην συνεδρίαση μετά την, που θα ακολουθήσει μετά την υποβολή του εγγράφου, του σχεδίου εγγράφου από το Συμβούλιο. Κύριε Κόπμαν, σας ευχαριστούμε για την παρουσίαση αυτή. Σας ευχαριστούμε για τη συζήτηση. Ολοκληρώνεται κατά αυτόν τον τρόπο η πρωινή μα συνεδρίαση και θα συνεχίσουμε με την απογευματινή μας συνεδρίαση στις 3 το μεσημέρι. Σας ευχαριστώ.